23 με 26 που γίνεται. Το θέμα είναι για το πώς θα εμποδίσουμε τη βία. Ένα θέμα για το οποίο εμείς, ε, μας είναι προσφυλές στην Επιτροπή μας. Θεμελιώδες θέμα θα έλεγα για τα δικαιώματα των γυναικών. Γυναίκες που ζουν υπό το κράτος του φόβου φοβούμενες την κακοποίηση. Φοβούνται για τη ζωή τους. Τέτοιες γυναίκες πραγματικά δεν μπορούν να λάβουν μέρος ούτε στον χώρο, στην εργασιακό χώρο, ούτε στο κοινωνικό. Ενώ αυτό αποτελεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ξέρουμε πόσο, πόσο μεγάλη έκταση έχει αυτή η βία. Μιλάμε τώρα για σωματική, ψυχική βία κτλ. Και είναι πολλές, πολλές διεθνείς οργανώσεις και τα Ηνωμένα Έθνη που δουλεύουν με πολλούς τρόπους για να μπορέσουμε ε, να καταπολεμήσουμε αυτή την πληγή θα λέγαμε, τη βία κατά το γυναικών. Επίσης να πω ότι έχει γίνει μια μεγάλη εκστρατεία με το θέμα «Πες όχι στη βία κατά των γυναικών». Και αυτό έχει υποστηριχθεί από ανθρώπους από πολλές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη στράτευση ε, σε αυτόν τον αγώνα. και θα επίσης μπορεί να ξεκινήσει κανείς και με άλλα ε, με άλλη μέσα σε αυτή την εκστρατεία. Και σίγουρα η Επιτροπή μας έχει μια μεγάλη ευθύνη για να δουλέψουμε, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βία που πλήττει τις γυναίκες είναι κάτι το οποίο είναι ε, εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμποδίζει τη συμμετοχή μας, ε, των γυναικών δηλαδή, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Μια μικρή λοιπόν εισαγωγή για το ψήφισμα, το κείμενο αυτό. Όλοι το έχετε στη διάθεσή σας και να εκφράσετε, θα ήταν καλό, τις απόψεις σας για να περάσουμε στην ψηφορία. Αυτό αποτέλεσε λοιπόν μια μικρή εισαγωγή για να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να δουλεύουμε με αυτό το ψήφισμα και να έχουμε ένα διάλογο στην ε, Ολομέλεια για να συνεχίσουμε το έργο μας πάνω σε αυτό το τομέα. Οι συνάδελφοι μπορούν να πάρουν τώρα το λόγο για να εκφράσουν απόψεις επί του κειμένου ψηφίσματος, το οποίο είναι, διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Ματέρα. Λοιπόν, ανέλησα τις 73 τροπολογίες που παρουσιάστηκαν για το ψήφισμα και διαπίστωσα ότι πολλές από αυτές τις έννοιες επαναλαμβάνονται και δεν προσθέτουν και κάτι ε, επιπλέον. Αντιθέτως βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες κάποιες τροπολογίες ε, συναδέλφων, τις οποίες προσωπικά αποφάσισα να διατηρήσω ενώ και εγώ έκανα λίγες ε, τροπολογίες με κάποιες νέες ε, έννοιες. Προσπάθησα να αποφύγω πολλές επαναλήψεις. Στόχος μου ήταν η απλούστευση διότι διαπίστωσε και από τον όγκο των τροπολογιών που προέκυψαν ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλες. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο και στο οποίο ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Ελπίζω λοιπόν αυτό που θα κάνουμε σήμερα ε, να οδηγήσει σε ένα σημαντικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη όθηση σε ε, πρωτοβουλίες ακριβώς για αυτό το θέμα, διότι όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για την προσοχή που έδωσε όλη η Επιτροπή ε, στο θέμα αυτό. Εύχομαι λοιπόν καλή δουλειά σε όλους και να συνεχίσουμε πάντα έτσι. Ευχαριστούμε την κυρία Ματέρα. Άλλος, άλλη. Αν όχι, τότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Και ζητώ, α, κυρία Παβανόβα, αλλά να πω πρώτα ότι συνάδελφοι, συναδέλφισες, για βγάλτε την κάρτα σας να τις έχουμε στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Κυρία Παβανόβα. Thank you, Madam Chair, giving the fact that... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή κάποιοι από τους συναδέλφους μας ε, σε μία ώρα πρέπει να φύγουν γιατί πρέπει να πάνε στη Μαδρίτη για την ε, επίσκεψη αντιπροσωπείας, έχω να πω το εξής, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για την τροπολογία 59. Στο αγγλικό κείμενο, είναι μια γλωσσική παρατηρήση, στο αγγλικό κείμενο γράφουμε ότι γυναίκες που είναι θύματα βιασμού θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια. Στη βουλγαρική εκδοχή λέει δωρεάν νομική βοήθεια. Το πρωτότυπο είναι τα ισπανικά. Ισχύει το δωρεάν νομική υποστήριξη που έχω στη βουλγαρική εκδοχή. Νομίζω ότι είναι ακόμη προτιμότερο να είναι δωρεάν η νομική υποστήριξη. Κυρία Παβανόβα, θα το δούμε αυτό το γλωσσικό που θίξατε. Ναι, μου λένε ότι είναι free, free. Είναι σαφέστατα για το ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ξεκινάμε για την ψηφοφορία μας. Και θα ξαναπροσπαθήσω με τα αγγλικά, δίνοντας τον, τους αριθμούς τροπολογιών ε, για να προχωρήσουμε. Αν δεν λειτουργήσει τα πράγματα, θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τροπολογία 31, χωρισμένη σε 7 διαφορετικά τμήματα. Επομένως, θα, ψηφίσουμε πρώτα το τμήμα 1, υπέρ, τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τμήμα Τροπολογία λοιπόν 31 ε, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς ε, το τμήμα 1 πέραση ψηφοφορίας 9 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Επομένως απορρίπτεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα 3. Υπέρ. Καταπίπτει. Συγγνώμη. Άρα μπορούμε να περάσουμε στην ε, τροπολογία 32 υπέρ τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 35 η οποία μπορεί να συνδυαστεί με την 34 και την 36 πρέπει να τις ψηφίσουμε όμως ξεχωριστά. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, ε, δούλεψε τώρα. Εκτός ε, μικροφώνου το σχόλιο. Okay. The vote is closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. 8 ψήφοι υπέρ, 13 κατά και 2 αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 41 καταπίπτει και περνάμε στη 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 45 είναι σε δύο τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 καταπίπτει. Ψηφίζουμε το τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. για το δεύτερο τμήμα της 46. Πέρας της ψηφοφορίας. 11 ψήφοι υπέρ, 16 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49, ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 51. Καταπίπτει και αυτή. Περνάμε στην 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία. Για την τροπολογία υπαριθμών 53. Πέραση της ψηφοφορίας. 16 ψήφοι υπέρ, 11 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Δεν χρειάζεται να ελέγξουμε νομίζω. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας έχουμε 16 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 ψήφους υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Για την 68 ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει. Τέλος της ψηφοφορίας. 12 ψήφοι υπέρ, 15 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Τέλος της ψηφοφορίας. 11 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Α, είναι ταυτόσιμες με την 10 και την 11 ψηφίζουμε λοιπόν ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όλες δηλαδή εγκρίνονται ή να το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την 9 και 10 και 11 9 και 10 διορθώνω 9 τροπολογίες 9 και 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά και 2 αποχές. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 αποσύρεται. Περνάμε στην 16 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε για τη 16? Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Πέραση της ψηφοφορίας. 14 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάσαμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρόεδρε, ίσως να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι στην πρώτη παράγραφο αν απορρίπτονται τα πρώτα δύο τμήματα θα πρέπει να ψηφίσουμε για τα υπόλοιπα δύο, αλλά δεν τα ψηφίσαμε. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε πώς έχει η κατάσταση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Κοιτάξτε, το πρώτο και το δεύτερο μέρος απορριφθήκανε. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα μέρη είναι εκτός νοήματος από τη στιγμή που απορριφθήκαν το πρώτο και το δεύτερο μέρος. Γι' αυτό δεν υπήρχε λόγος να ψηφίσουμε, καταλάβατε. Ωραία. Πάμε για την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. η ομάδα των σοσιαλιστών έχουν ένα άτομο παραπάνω στην ψηφοφορία εδώ. εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πέρασε ψηφορία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πώς ψηφίσετε. Ναι ή όχι. Κατά, κατά. Εντάξει. Θα βάλουμε στα κατά άλλη μία ψήφο. Λοιπόν, έχουμε 17 υπέρ του ψηφίσματος, τρεις κατά, τέσσερις δηλαδή με την κυρία Λούλη και είχαμε και τέσσερις αποχές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για αυτήν εδώ την ψηφοφορία και για το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. Προτείνω να ξαναρχίσουμε λοιπόν, να συνεχίσουμε μάλλον το έργο μας. Το σημείο που έχουμε τώρα είναι ενημέρωση μετά τη συνάντηση των συντονιστών που είχαμε νωρίτερα, τρεις με τέσσερις, εμείς είχαμε τη μια σειρά εκθέσεων τροπολογιών, ε, τρο, ε, ε, εκθέσεων πρωτοβουλίας και η Γκουε ανέλαβε το θέμα του δικού χάρτη για την ο, ισότητα, οι πράσινοι ανέλαβαν την έκθεση πρωτοβουλίας για τα θέματα, τις πτυχές της ισότητας όσον αφορά την οικονομική κρίση μετά έχουμε αυτή που έχει να κάνει με τη θέση των γυναικών σε ηγετικέ θέσεις. Είναι το ΕΛΚ που την έχει αναλάβει αυτή την έκθεση πρωτοβουλία και η Άλντε είναι το θέμα που έχει να κάνει με την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών που ανήκουν σε διάφορες εθ... μειονότητες εθνικές. Αποφασίσαμε αν η Επιτροπή Περιβάλλοντος κάνει δική της έκθεση όσον αφορά την αλληλεγγύη και την υγεία και για το ΠΕΣ θα μειώσουμε τα, τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε μια γνωμοδότηση εμείς. Αποφασίσαμε ότι η κυρία Μπάουερ θα αναλάβει αυτή θα αναλάβει όσον αφορά το οικονομικό έτος του 2008. Επίσης πήραμε την απόφαση για αναφορές που γίνανε εδώ στην Επιτροπή και όλοι θα ενημερώνονται, όλες οι συναδέλφες θα ενημερώνονται για αυτές τις αναφορές. Επίσης, έχουμε ένα, έχουμε ένα θέμα από την κυρία Μαρκαντίνη που αφορά τις μουσουλμάνες γυναίκες στην Ευρώπη και το θέμα της Μπούρκα, τη χρήση της Μπούρκα, ε, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα ενημερώσει ο πρόεδρος το άτομο το οποίο έχει θέσει αυτή την ε, ερώτηση. Επίσης, άλλο ένα θέμα για αναφορές που και αυτό δεν, αφορού, δεν ήταν στα πλαίσια της εντολής μας, και πάνω σε αυτό θα ενημερώσουμε όλα τα μέλη. Επίσης μια άλλη απόφαση ότι θα υπάρξει ένα ψήφισμα για τη διεύρυνση για προς την Μακεδονία, την Τουρκία και την Κροατία και αποφασίσαμε να συμβάλλουμε σε αυτό το ψήφισμα μέσω παραγραφών οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Επίσης, ε, αποφασίσαμε για το χρονοδιάγραμμα, για ακροάσεις, αντιπροσωπίες και η γραμματεία φυσικά θα σας ενημερώσει, θα ενημερώσει όλες, όλα τα μέλη για αυτές τις ε, ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί. Ακόμα ένα θέμα είχε να κάνει με την ακρόαση για ποια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά την ισότητα. Αποφασίσαμε για μια προθεσμία, 13 Νοεμβρίου, οπότε όλες οι πολιτικές ομάδες θα μας ενημερώσουν για το πώς βλέπουν ε, για ε, την οργάνωση αυτής της ακροάσεως. Και τέλος, αποφασίσαμε όσον αφορά όσον αφορά τις ακροάσεις μας για τα μέλη που θα προτείνονται είχαμε συζητήσει και το πρωί ότι ε, όσον αφορά τις ακροάσεις με τους επιτρόπους ε, εκφραστήκαν κάποιες απόψεις τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε στους προτινόμενους και εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι οι προτάσεις μας αυτές θα σταλούν σε όλα τα μέλη. Οι συντονιστές συμφωνήσανε ότι ε, χρειαζόταν η περαιτέρω ε, προτάσεις όπως διαμορφώθηκε αυτό κατά τη διάρκεια της πρωινή συνεδριάσεως και τέλος τέλος αποφασίσανε οι συντονιστές επίσης ότι όσον αφορά τους ε, επιτρόπους τα διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία θα προταθούν εμείς από τη δική μας ε, επιτροπή να γράψουμε μια επιστολή προς τον πρόεδρο και να εκφράσουμε επιθυμίες λέγοντας ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένας επίτροπος ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα ε, το θέμα της ισότητας. Αυτά εμπεριλήψει από τη συνάντηση των συντονιστών και φυσικά θα ενημερωθούν όλα τα μέλη για ε, αυτό, για αυτές τις αποφάσεις. Έχουμε κάποια θέματα ακόμα στην ημερήσια διάταξη. Εγώ θα σας αφήσω όμως. Υπάρχει μια αντιπροσωπεία που θα πάει στη Μαδρίτη σήμερα και χαίρομαι που η κυρία Εστρέλα που δέχτηκε να συνεχίσει, να αναλάβει μάλλον την Προεδρία για το υπόλοιπο της ε, ημέρας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη σημερινή μας συνεργασία και παραδίδω την σφύρα του του Προέδρου στην ε, συνάδελφο Εστρέλα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αλλά έριχνα μια ματιά στην ημερήσια διάταξη για να δω τι μας έχει απομείνει. πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων. Η, η, κυρία, η συντάκτρια συγγνώμη, η κυρία Μπάουερ και της δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους όσους είναι παρόντες, καταρχάς. Είμαι βέβαιη ότι για κάποιους από εσά θα είναι έκπληξη να έχουμε αντί για γνωμοδότηση ή σχέδιο γνωμοδότησης μια προφορική ερώτηση. Ξέρετε ότι αυτό προέκυψε και από τη νέα θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την υπογραφή της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, από τον τελευταίο πρόεδρο. Προσπαθούμε λοιπόν να, προσλα... να προλάβουμε να τελειώσουμε το θέμα αυτό πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, η μόνη δυνατότητα να αποστείλουμε ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε και αυτό που περιμένουμε από αυτούς είναι να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση μαζί με ψήφισμα. Η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξή. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή την άγουσα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πλέον δύο προφορικές ερωτήσεις. Η μία βέβαια απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η άλλη στο Συμβούλιο. Αλλά έχουμε και δύο διαφορετικές εκδοχές, διότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, ετοίμασε μία διαφορετική εκδοχή της προφορικής ερώτησης και θα πρέπει μαζί με την κυρία Χέντ, η οποία είναι συντάκτρια της προφορικής ερώτησης, να ετοιμάσουμε μια κοινή εκδοχή και ε, για την προφορική ερώτηση αλλά και για το ψήφισμα. Πιστεύω ότι θα έχουμε χρόνο να επανέλθουμε στο θέμα και θα έχουμε μια κοινή εκδοχή. Θεωρείς ότι σήμερα απλά έχουμε μία άτυπη ανταλλαγή απόψεων για να δούμε λίγο τι θα θέλαμε να έχουμε στο κοινό κείμενο με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ σε αυτή τη φάση είναι ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα αυτό και ναι, μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας ετοιμάσει μια νέα εκδοχή, κατά πάσα πιθανότητα όμως θα είναι αντίστοιχη με αυτήν που θα εγκρίνει το Συμβούλιο κάπου προς τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου Και αυτή είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως να είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο όσο περιμέναμε, αλλά θα είναι πολύ μεγάλο. Αν θυμάστε, κάναμε τεράστια προσπάθεια με το θέμα των ε, παιδιών που ε, ζητιανεύουν στους δρόμους μεγάλων πρωτευουσών κρατών μελών. Πολλά από αυτά τα παιδιά όπως μας είπε και η Europol, είναι θύματα εμπορίου. Ορισμένες φορές, ακόμα και με τις μητέρες τους ή με ολόκληρες οικογένειες. Και δεν είχαμε κανένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, διότι ήταν ανέφικτο να προσκομίσουμε οποιαδήποτε απο, ε, απόδειξη και επειδή η διακονία δεν είναι παράνομη βάσει των ε, νομικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρχε στην πράξη κανένα μέσο στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το έγκλημα και να το θεωρήσουμε αδίκημα που έχει να κάνει με την εμπορία ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή κατατάσσεται σε ένα κατάλογο και θεωρείται μια ακόμα μορφή εμπορίας. Στα πλαίσια λοιπόν της προστασίας των θυμάτων προσπαθούμε να ε, μην έχουμε περιπτώσεις στις οποίες ε, έχουμε επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και τα θύματα ε, ξαναπέφτουν στην ίδια παγίδα Φυσικά θα υπάρχει και κάποιος, ε, κάποια δυνατότητα να ε, συζητηθεί και η δική μας η πρόταση, διότι ε, εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχουν δωρεάν νομικές συμβουλές για τα θύματα. Στο, δεν υπάρχει αυτό το θέμα στο σχέδιο κειμένου. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα προσαγωγή σε δίκη ακόμα και διαμεθοριακά, αλλά όχι για κατοίκους τρίτων χωρών, μόνο για ε, υπηκόους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα της προστασίας των παιδιών και όσον αφορά τις κυρώσεις ε, δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να ελέγξουμε ίσως αργότερα όταν θα έχουμε και ένα σχέδιο κειμένου είναι η σοβαρότητα των κυρώσεων. Πέρσι είχαμε μια αξιολόγηση αντικτύπου η οποία κατέδειξε ότι σε κάποιες χώρες οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ ήπιες ε, υπέρ το δέον. Ε, βέβαια όταν αρχίσαμε να συζητάμε το θέμα της εμπορίας ανθρώπων υπήρχε και κάποιο κράτος μέλος όπου μπορούσε κάποιος να τιμωρηθεί απλά και μόνο με ένα πρόστιμο. Βέβαια η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει μετά από το τελευταίο πλαίσιο και το τελευταίο πρόγραμμα δράσης. Να συνοψίσω όμως, η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο σχέδιο προφορικής ερώτησης. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το κείμενο και θα συνεχίσει φυσικά και η επεξεργασία του ψηφίσματος. Δυστυχώς η κυρία Χέντ αυτή την εβδομάδα δεν είναι εδώ. Γι' αυτό και το θέμα ε, έχει παρεπευθεί στο Δεκέμβριο και κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπάουερ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι να ζητούν το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Έρνστ. Κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Ήθελα να σχολιάσω το θέμα αυτό γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι το να έχουμε επακριβείς διατυπώσεις ακριβώς για αυτό το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων που είναι μια έννοια πολύ ευαίσθητη και θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς πώς θα δώσουμε τους ορισμούς και θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δεύτερον, για τις πιο αυστηρές ποινές θα πρέπει να δούμε και στα κράτη-μέλη τι ισχύει σε κάθε περίπτωση και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ συγκεκριμένα πού θέλουμε να έχουμε πιο αυστηρές ποινές γιατί μερικές φορές μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές οι πιο αυστηρές ποινές και όταν μιλάμε ε, για παιδιά ως θύματα ε, μπορεί να είναι ε, και πιο προβληματικές οι πιο αυστηρές ποινές Τα λέω αυτά από την οπτική γωνία τη Γερμανία. Μπορεί κάποιε άλλε χώρε να το βλέπουν διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει πολύ συγκεκριμένα να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι ε, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι πρέπει ε, να τονίσουμε την προστασία των θυμάτων. Και όσον αφορά τα παιδιά, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Υπάρχουν διάφορες ε, μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν όταν ε, τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες, παραδείγματος χάρη, όταν ε, είναι θύματα. Θα ήθελα να πω ότι είναι θετικό ότι ασχολείται με τα θέματα αυτά η κυρία Μπάουερ. Θεωρώ πολύ σωστό να προχωρήσουμε με τον τρόπο που προτείνεται και ευχαρίστω να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή. Παρακαλώ όμως να μας δοθεί δυνατότητα να εξετάσουμε πολύ συγκεκριμένα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να δούμε και τι σχέσεις ε, μπορεί να υπάρχουν ε, και με οργανισμούς όπως η Frontex. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν ανεξέλεγκτο οργανισμό και γι' αυτό ε, νομίζω ότι πρέπει πολύ συγκεκριμένα να εξετάσουμε το πώς θα προχωρήσουμε, να δούμε και το χρονοδιάγραμμά μας. Και αυτά είναι θέματα που για την ΓΚΟΕ είναι πολύ σημαντικά. Υποστηρίζουμε και εμείς αυτά τα θέματα που ανέφερε η κυρία Μπάουερ και άλλοι συνάδελφοι. Είναι ερωτήματα που πρέπει να τεθούν και θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα. και με την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας νομίζω ότι θα αλλάξουν πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστούμε, κυρία Έρνστ. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ το θεωρώ πολύ θετικό το ότι στην Επιτροπή μας ε, μπορούμε να εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Και θα ήθελα να σχολιάσω ένα συγκεκριμένο σημείο, το 6α, για αυτούς που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ε, που έχουν σχέση ε, με ε, θύματα εμπορίας. Και ας μην ξεχνάμε και την περίοδο που είχαμε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Γερμανία υπήρξαν θέματα που συζητήθηκαν πάρα πολύ και χρειάζεται επεξήγηση δεν μπορούσαμε να εμποδίσουμε κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων ποδοσφαίρου την εκμετάλλευση των θυμάτων και ξέραμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες αυτών των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ε, και έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να πληροφορήσουμε και να ενημερώσουμε και αυτούς που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. Γι' αυτό για το σημείο 6α νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε γιατί είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ναι, θυμόμαστε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του πρωταθμίωτος ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Και έχουμε αναλάβει δραστηριότητες και συνεργαστήκαμε και με τις γερμανικές αρχές και όλα αυτά συνεισέφεραν στο να αποφύγουμε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Άρα νομίζω ότι ήταν θετικά τα αποτελέσματα των εργασιών μας. Κυρία Κώστα. Καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Μπάουερ για τη συνεισφορά της ε, επειδή ξαναείδαμε λίγο για τη διαδικασία και αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε την προφορική ερώτηση για να παρουσιάσουμε τη θέση μας, ουσιαστικά νομίζω ότι είναι η πρώτη επίσημη πράξη που κάνουμε ως Επιτροπή ε, λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να δράσουμε με μια άλλη διαδικασία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή μας μαζί με το Κοινοβούλιο, μαζί και με την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ θέλει να συνεχίσει να εργάζεται για να ενημερώσουμε το πλαίσιο του 2002. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά τα διάφορα ερωτηματικά που παρουσιάζονται. Μου φαίνεται ότι το σημείο 6β είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το θέμα δηλαδή της συνένεσης και το γεγονός ότι δεν Να σας το πω αλλιώς. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιες φορές να συνενέσει ένα θύμα είναι τέτοιος ώστε ε, μπορεί να είναι θύμα εμπορίας παρά το γεγονός ότι φαινομενικά φαίνεται να συνενεί σε κάτι. Ε, πολύ συχνά διαπιστώνουμε σήμερα ότι κάποια άτομα είναι σε ευάλωτη θέση και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και θα πρέπει λοιπόν αυτό να θεωρείται πάντα αδίκημα εμπορίας ε, αν και ε, κατά τα φαινόμενα μπορεί να μην υπάρχει σωματική βία αλλά υπάρχει κάποια μορφής πίεση. Πολλές φορές διαπιστώνουμε στη χώρα μας, ε, τουλάχιστον στην Ιταλία αυτό συμβαίνει, ότι αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εμπορία ανθρώπων. Όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό ε, το 1996 είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Λευκή Βίβλο για την εμπορία ανθρώπων και από εκεί και πέρα υπήρξε και σχετική νομοθεσία από τα κράτη-μέλη και ε, γινόταν αναφορά σε μία πολύ ε, προφανή κατάδειξη της σωματοπορίας. Ε, σήμερα το οργανωμένο όγκλημα ε, προσαρμόστηκε στους πιο αυστηρούς κανόνες που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Τα άτομα τα οποία είναι θύματα πολύ συχνά είναι σε σπίτια, δεν βρίσκονται στους δρόμους, είναι πιο αόρατα αν θέλετε. Δεν μπορούμε πάντα να εντοπίσουμε πού ακριβώς ε, έχουμε εμπορία απονομικής τουλάχιστον σκοπιάς και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν τα μέτρα που ε, παραδοσιακά λαμβάνονταν. Ε, ίσως εγώ ως νέα δεν τα γνωρίζω καλά. Θα ήθελα να ξέρω αν παρουσιάστηκε η έρευνα για την κατάσταση της εμπορίας ανθρώπων που έπρεπε να είχε παρουσιαστεί ε, ήδη το φθινόπωρο του 2009, διότι ξέρω ότι από όλα τα κράτη-μέλη ζητήθηκε να γίνει μια κάποια έρευνα ώστε να υπάρχει μια παρακολούθηση της κατάστασης που έχει αλλάξει σε σχέση με κάποια χρόνια πριν. Αυτή λοιπόν η προσαρμογή δυστυχώς ε, των ε, εγκληματικών οργανώσεων στους πιο αυστηρούς νόμους παραδόξως είναι ένα επιπλέον πρόσκομα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ακόμα και αυτά που προβλέπονταν το 2002. Αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε λοιπόν και αυτή την ησυχία στο κείμενο της ερώτησης, ε, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, διότι νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα διαπιστώνουν και πολλές αστυνομικές ε, ε, δυνάμεις. Φαίνεται ότι πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι εμπορία. Υπάρχει μια συνένεση και δεν φαίνεται να είναι βεβαιασμένη όλη αυτή η διαδικασία. Ε, είναι κάτι το οποίο ε, διαπιστώνουμε και στη χώρα μας παρά το γεγονός ότι έχει εγκρίνει πριν από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νομοθεσία υπέρ των θυμάτων. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Κυρία Μπάουερ, θέλετε να παρέμβετε για να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Φυσικά. Ε, καταρχήν θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ενδιαφέρουσα ιστορία την άκουσα στη Βιέννη σε μια διάσκεψη για τη μετανάστευση. Μας έδειξε κάποιος μια φωτογραφία που βλέπουμε ένα τασάκι με μια επιγραφή που έλεγε να σταματήσουμε την εμπορία κοριτσιών και η ημερομηνία ήταν 1909. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η εμπορία ανθρώπων ε, εκείνη την εποχή ήταν εμπορία κοριτσιών από την Ευρώπη, μεταξύ Ευρώπης ε, και Λατινικής Αμερικής. Θέλω να πω ότι δεν είναι καινούρια υπόθεση η εμπορία ανθρώπων, είναι μια παλιά ιστορία και βλέπουμε πόσο διαρκεί αυτή η παλιά ιστορία. Μερικές φορές βλέπουμε ότι η αστυνομία λειτουργεί σωστά. Βλέπουμε ότι μερικές φορές τα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται καλά. Μπορούν να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, αλλά εδώ χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία που δεν λειτουργεί πάντοτε. Χρειαζόμαστε εδώ διεθνή συνεργασία μεταξύ της Frontex, της Eurojust, της Europol, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, πράγμα το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εμφανώς εδώ πρόκειται για ένα θέμα πολύπλοκο. Και πρέπει να δούμε ε, τι μπορούμε να πούμε για να καλύψουμε τα σημαντικότερα θέματα. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε σελίδες επί σελίδων χωρίς ε, να είναι σημαντικά αυτά τα οποία λέμε σε κάθε γραμμή της κάθε σελίδας. Και μία συμφωνία πλαίσιο που θα μπορούσε να είναι η κατάληξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Καταρχήν το θέμα των ορισμών. Υπάρχουν πολλοί καλοί ορισμοί και αλλάζουν αυτοί οι ορισμοί. Υπάρχει το πρωτόκολλο του Παλέρμο που ορίζεται η εμπορία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης έχει μία σύμβαση με έναν ορισμό και η συμφωνία πλαίσιο επίσης περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό ορισμό. Υπήρχε, σε ένα προηγούμενο, υπήρχε ένας προηγούμενος ορισμός που δεν περιλάμβανε την ε, εμπορία οργάνων. Τώρα έχουμε και τον ε, ορισμό που συμπεριλαμβάνει την εμπορία οργάνων για το Συμβουλίο της Ευρώπης. Υπάρχουν δηλαδή πολλά διαφορετικά όργανα και δημιουργείται σύγχυση με τους διαφορετικούς ορισμούς που υπάρχουν. Και υπάρχει και διαφορά μεταξύ εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίου ανθρώπων. Υπάρχουν ε, στοιχεία που μας επιτρέπουν στο τέλος της διαδρομής αυτών των ανθρώπων να κρίνουμε αν πρόκειται για εμπορία ή για λαθρεμπόριο ανθρώπων, αν έχουν πληρώσει χρήματα για να μεταφερθούν κάπου ή αν ε, μεταφέρονται ως θύματα. Τώρα όσον αφορά την προστασία των παιδιών, ε, ήθελα να προσθέσω κάτι, πολύ σωστά το τόνισε η κυρία Έρνστ δεν πρέπει να τιμωρούνται τα θύματα, ακόμη και αν τα ίδια τα θύματα διαπράττουν αξιόπινες πράξεις. Και στη συμφωνία πλαίσιο νομίζω ότι ακολουθούμε πολύ προσεκτική διατύπωση. Ιδίως όταν εμπλέκονται παιδιά. Όταν γίνεται εξέταση παιδιών ε, ε, ως μαρτύρων ε, λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα γίνεται αυτό. Και στο σημείο 6β επίσης προσφέρεται μια σημαντική ευκαιρία γιατί ξέρουμε ότι λειτουργεί δυστυχώς και το σύνδρομο της Στοκχόλμης που κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και ξέρουμε ότι με μια συμφωνία πλαίσιο δεν μπορούμε να επιτύχουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύησεις για τα πάντα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να κάνουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας για να επιτύχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Σαφώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα. Δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα και είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας από 1η Δεκεμβρίου ελπίζουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μπορούμε ε, να ασχοληθούμε και με αυτό το τομέα εντατικότερα και θα έχουμε και το δικαίωμα συναπόφασης. Ακούσαμε λοιπόν πολλά σχόλια. Νομίζω ότι συμφωνούμε επί της διαδικασίας που πρότεινε η κυρία Μπάουερ. Θα κάνουμε μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και επιπροσθέτως θα συντάξουμε και ένα σχέδιο ψηφίσματος. Θα μπορούσε η κυρία Μπάουερ να είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, θα μπορέσουν να συνεργαστούν και οι ισχυώδεις εισηγητές και αυτό το ψήφισμα θα μπορέσουμε να το εγκρίνουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 30 Νοεμβρίου, στις 3 το απόγευμα. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος λοιπόν θα μπορέσει να συζητηθεί σε εκείνη τη συνεδρίασή μας και στη συνέχεια να συζητηθεί στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο 14 έως 16 Δεκεμβρίου. Αυτά λοιπόν και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους εσάς που συμμετέσχετε και τους διερμηνείς. Ευχαριστή η Πρόεδρος, που όπως πάντοτε ήταν πολύ αποτελεσματική. Και οι διερμηνείς ευχαριστούν την Πρόεδρο για τα καλά της λόγια.